Ε, Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα ένα αίτημα. παρέμβαση από τον κύριο Πόσπης. Λέγεται το λόγο. Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο κόσμος να μάθει περισσότερο αυτές τις αξίες και από την τσεχική εμπειρία γνωρίζω ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις αξίες ε, στα πλαίσια της παιδείας και έτσι να μαθαίνουν αυτές τις αξίες οι νέοι, γιατί πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν περί τίνος τι είναι ευρωπαϊκέ. υπό την ε, επίρρεια της παραπληροφόρησης δεν καταλαβαίνουν ότι η Ένωση είναι μια ελεύθερη ένωση χωρών που είναι υπέρ δικαιωμάτων, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Πολλές φορές κάνω περιοδίες στα σχολεία και εντυπωσιάζομαι από την άγνοια των νέων σε σχέση με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ θετική την αύξηση της χρηματοδότησης για αυτό το πρόγραμμα. Πολύ καλό είναι. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Και έτσι εδώ ολοκληρώνεται το κατσδιά και θα δώσουμε το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η συζήτηση αυτή δείχνει τη σημασία που δίνουμε στην προαγωγή των δικαιωμάτων και αξιών και η υποστήριξη για το πρόγραμμα το οποίο προτείνει η Επιτροπή για το Μέλλον δείχνει πόσο σημαντικό είναι. Είναι ε, πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τις διαφορετικές ερμηνείες του τι σημαίνει η λέξη ισότητα. Μπορώ να σας εξομολογηθώ ως Επίτροπος υπεύθυνη για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη ότι όταν ήρθα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσα ότι πρέπει να προωθούμε την ισότητα. Εγώ έζησα τη μισή ζωή μου σε ένα καθεστώς που επέβαλε την ισότητα. Ισότητα υπό την έννοια που ανέφερε η κυρία Σόντροβα, δηλαδή υπό την έννοια της ομοιομορφίας. Ζούσα σε μια κοινωνία όπου δεν βλέπαμε τους ανθρώπους σε αναπηρικά καροτσάκια. Ζούσα σε μια κοινωνία όπου δεν θυμάμαι να είδα ποτέ μου κάποιο άτομα με ψυχικές νόσους γιατί τους έκρυβαν. Τους έκρυβαν για να μην τους βλέπει ο κόσμος γιατί δεν ήταν ιδανικοί με τους υπόλοιπους εντός εισαγωγικών ίσους σοσιαλιστές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διευκρινίσω ότι μιλάμε για ισότητα έναντι του νόμου. Μιλάμε για την αρχή του ότι όλοι έχουν τα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και έχουμε και καθήκον να προστατεύουμε τους αδυνάμους καταπολεμώντας κάθε μορφή διάκρισης. Ταυτόχρονα, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι προωθούμε την πολυμορφία τον πλουραλισμό, το διάλογο, τη δραστηριοποίηση των πολιτών. Και όταν μιλώ για διάλογο, γνωρίζετε ότι είμαι υπεύθυνη και για την ισότητα των φύλων. Προσπαθώ να υλοποιήσουμε την ε, επικύρωση της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις εκκλησίες και ζήτησα από τις εκκλησίες να προσέλθουν σε διάλογο γιατί θέλω να ακούσω τα επιχειρήματά τους. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να ακούσουμε διστάμενες απόψεις. Και δεν νομίζω ότι κανείς εδώ θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια για να μην αφήσει να μιλήσει κάποιος που έχει διαφορετική άποψη. Και βέβαια υπάρχουν κάποια όρια για την ελευθερία της έκφρασης. Μπορεί κάποιοι από εσά να λέτε ότι σε κάποιους επιβάλλουμε τη σιωπή. Ναι, θα επιβάλλουμε τη σιωπή σε αυτούς που είναι υπέρ της βίας και της δολοφονίας άλλων. Και στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Και γι' αυτό ζητάμε από τις ε, εταιρείες να διαγράφουν μηνύματα μίσους, ε, μηνύματα που μπορεί να προάγουν τη βία στην καθημερινή ζωή. Ζητάμε από τις εταιρείες να διαγράφουν τέτοια μηνύματα. Δεν θέλουμε ελευθερία έκφρασης για, αυτούν, αυτούς που θέλουν να διαπράξουν εγκλήματα. Προάγουμε τον διάλογο, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες με κριτική σκέψη να αποφασίζουν τι είναι σωστό και τι πρέπει να ανέχονται. Όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι ενεργοί πολίτες προσδιορίζουν το τι είναι ανεκτό. Γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες, ένα πρόγραμμα που ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί με έξυπνο τρόπο για να βοηθήσει την κοινωνία να αυξήσει την ανεκτικότητα και την κατανόηση μεταξύ όλων, ούτε ώστε να υπάρξει η διαφοροποίηση και η πολυμορφία. θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε την κοινωνία να ευημερεί και το διάλογο των πολιτών ε, να ανθίσει. Ανέφερα τον τομέα του διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και του διαλόγου. Πάντοτε είμαι υπέρ της προαγωγής της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας μας. Αλλά όπως γνωρίζουμε και καταχρήσεις υπάρχουν στον τομέα του διαδικτύου. Με ρητορική μίσους, ε, προάγοντας επιθέσεις κατά πολιτών. Ε, τέλη Ιανουαρίου θα πάρω την έκθεση από τις εταιρείες πληροφορικής με στοιχεία για ένα χάρτη μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας κατάλογος των συνήθων υπόπτων στον κατάλογο αυτών που προάγουν το μίσος. Έχουν τις μειονότητες, έχουν τις εκκλησίες, άτομα που εκφράζουν ανοιχτά τις θρησκευτικέ τους απόψεις, συμπεριλαμβανομένων και χριστιανών, τους ομοφιλόφιλους, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς σε πολλές χώρες και τους δικαστές. Όλους αυτούς συμπεριλαμβάνουν στον κατάλογό τους αυτοί που προάγουν το μίσος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, γιατί πρέπει κάθε μέρα να θυμόμαστε ονόματα όπως ε, η Τζο Κόξ, ο Πάβελ Αντάμοβιτς, η Ντάφνε Καρουάνο Γκαλίσια, η Γιάν Μπούτσιακ. Και πολλοί ε, άλλοι μπορεί να γίνουν θύματα αυτού του μίσους. Αν δεν σταματήσουμε αυτή την τάση, φοβούμε ότι θα έχουμε και άλλα θύματα. Πώς να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κατάσταση. Μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση. Είμαι πεπισμένη ότι αν καταφέρουμε να προάγουμε την έννοια του ψηφιακού φόρου, φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τμήμα αυτών των κονδυλίων για την εκπαίδευση, όχι για προπαγάνδα, για εκπαίδευση για αντικειμενική πληροφόρηση για την ιστορία μας, για ενημέρωση της νέας γενιάς για να μπορέσει να αναπτύξει κριτικό πνεύμα, για να μπορέσει να επεξεργάζεται σωστά τις πληροφορίες. Και είμαι πεπισμένη ότι αν προάγουμε τις τεχνολογίες από τη μία πλευρά, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ωφέλη των τεχνολογιών και να χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό φόρο για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης και των αξιών για τις οποίες ε, συζητάμε. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Βαλέρο που είναι συγγήτρια. Για δύο λεπτά. I would like to, uh, you to put your headphone on. Ε, Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ε, όλους ε, όσοι εξέφρασαν την άποψή τους και επισήμαναν ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όταν μιλήσαμε για το πρόγραμμα αυτό. Ε, λάβαμε πολύ καλή τεχνική βοήθεια. Ε, Προσπάθησαμε να βρούμε λύση για τα προβλήματα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχω και κάποιες ανησυχίες. Είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι η Επίτροπος λέει ότι πράγματι ε, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, αλλά τελικά λένε ότι με λιγότερα μπορούν να κάνουν να πετύχουν ακόμα περισσότερα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή χρηματοδότηση για το σύνολο των προγραμμάτων. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν ε, τα προγράμματα λάβουν ε, μικρότερη χρηματοδότηση και χρειαζόμαστε και περισσότερα κονδύλια για τα νέα προγράμματα και τις νέες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το άρθρο υπαριθμών 2. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε πάρα πολλά ε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχουμε την επαρκή χρηματοδότηση. Ελπίζουμε αυτό να είναι δυνατόν. Ελπίζω να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ε, χρειαζόμαστε ικανοποιητικές δυτικά κονδύλια αλλά και οι νέοι τομείς θα πρέπει να διαχωρίζονται και να υποστηρίζονται. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αναφέρεται ότι αυτά θα μπορούσαν τα κονδύλια να αποκτηθούν ίσως από το Κοινωνικό Ταμείο και από αλλού, αλλά ε, σε τέτοιου είδους ε, ερωτήσεις, ε, σε κοινωνικά θέματα, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς από πού πρέπει να λάβει τα χρήματα. Κυρίως όταν πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. 13 εκατομμύρια ευρώ, αυτά είναι χρήματα που έρχονται από τις τσέπες των φορολογουμένων. Εδώ από ό,τι φαίνεται ε, πρόκειται για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε τα χρήματα για τα υφιστάμενα προγράμματα αλλά και για τα νέα προγράμματα. Νομίζω ότι είναι μια σαφή δήλωση αυτή και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλές συζητήσεις. Σύντομα θα αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να συμφωνήσουμε ε, παραδείγματος χάρη είναι, ε, ε, να αντιμετωπίσουμε μεγάλα θέματα και ελπίζω ότι θα έχουμε καλές και επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ε, ε, εισηγητές και τους ομιλητές ε, και την εισηγήτρια. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ευγενικό να κόβει κανεί να ε, παίρνει το λόγο από την εισηγήτρια. Γι' αυτό την άφησα να μιλήσει ενδεχομένω περισσότερο. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Ε, η πρώτη ανακοίνωση αφορά το ότι ο κύριος Μάικ Κούπεμ ε, πλέον ε, θα είναι στους μη εγγεγραμμένους από τον Ιανουάριο, 17 Ιανουαρίου του 2019. Και η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την ομάδα ESD για επιτροπές και αντιπροσωπείες αυτά μπορείτε να τα δείτε στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρξουν ε, τοποθετήσεις, αυτές οι αλλαγές θα θεωρηθούν ότι γίνονται δεκτές. Τώρα λοιπόν ε, έχουμε την ε, έκθεση της κυρίας Χάρμ σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης για την πάυση λειτουργίας του ποινικού εργαστήου Ιγναλίνα στην Λιθουανία. Και το λόγο έχει η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς για πέντε λεπτά. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, αξιότιμοι σκιοδησηγητέ, ε, κύριε Επίτροπε, ε, θα ήθελα για την περίπτωση που όλα αυτά που λέμε είναι ενδιαφέροντα για τη Λιθουανία. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τους πολίτες της Λιθουανίας, ε, κυρίως ε, τους πολίτες της περιοχής Γκυζικίνα. Ε, πήγα στην Γκυζικίνα, στην Λιθουανία, στο πυρηνικό εργοστάσιο Ιγναλίνα ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο το έχω επισκεφτεί τουλάχιστον 15 ε, φορές τα τελευταία χρόνια και έχω διαπιστώσει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση το να προτείνει ε, και να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις διαπραγματεύσεις με τη Λιτουανία το κλείσιμο αυτού του πυρηνικού σταθμού. Θέλω όμως να σας πω ότι εγώ μέχρι και σήμερα βρίσκω αυτή την απόφαση και σωστή και λογική. Διότι αυτό ε, ε, το ο πυρηνικός αντιδραστήρας ε, του τύπου RBMK1500. Αυτοί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Όσο λοιπόν ε, σημαντική ήταν αυτή η απόφαση για το, ε, την πάυση λειτουργίας του αντιδραστήρα, σωστή σας είπα για μένα αυτό. Ε, βέβαια οι Βρυξέλλες πίεσαν και αυτή η απόφαση συνδέθηκε με την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αφήσει όλο αυτό το κόστος στην Λιθουανία. Είναι ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας RBMK που κατασκευάστηκε ποτέ. Επιβλήθηκε από τη Μόσχα, αυτός ο αντιδραστής, στη Λιθουανία, που ήταν υπό την κατοχή της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι ισχυρίζονται οι Λιθουανοί. Σήμερα λοιπόν η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί ότι θα συμβάλλει στο κόστος και στο βάρος. Ε, και χαίρομαι που η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε μαζί μου το αρχικό ποσό που είχε προταθεί για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επταετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να μην παραμείνει ως έχει, αλλά να ε, αυξηθεί κατά 780 εκατομμύρια. Με αυτή λοιπόν την χρηματοδότηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το 26 ή πιο συγκεκριμένα το 27 θα είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί το μπλοκ 1 ή αν θέλετε και το μπλοκ 2 των δύο αντιδραστήρων. Σήμερα ε, θα αποφασίσουμε και αύριο θα ψηφίσουμε ε, για το ότι η σχέση ανάμεσα στην συμμετοχή της Λιθουανίας και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει ε, να παραμείνει η συμμετοχή ως προβλέπεται σήμερα. Η διαχείριση της ε, αποσυναρμολόγησης ε, στην Ιγκλαλίνα και πιστέψτε με, έχω πάει πολύ συχνά στην περιοχή αυτή. Αυτή η διαχείριση είναι σε πολύ καλά χέρια και αυτή είναι προϋπόθεση να υπάρχει σωστή διαχείριση της αποσυναρμολόγησης αλλά και μια διαφανής διαχείριση των οικονομικών. Και για αυτά υπάρχουν εγγύησεις, κατά τη δική μου άποψη. Η Λιθουανία εντωμεταξύ ε, με ένα δημοψήφισμα αποφάσισε ότι θέλει να εγκαταλείψει πλήρως την πυρηνική ενέργεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι σαφές για εμάς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό όχι μόνο πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά πιστεύω ότι η απόφαση που θα λάβουμε σήμερα για την αποσυναρμολόγηση και για την Ουγγναλίνα, αυτό θα πρέπει να συνδέεται και με το Όστρεβιτς στη Λευκορωσία, ε, που είναι πολύ κοντά στο Βίλνιο, σχεδόν φαίνεται σε τέτοια απόσταση. Ε, πρόκειται για ε, ένα πολύ επικίνδυνο πυρηνικό εργοστάσιο που είναι σχεδόν μάλιστα έτοιμο. Τα τεστ που έχουν γίνει για το Όστρεβιτς έδειξαν κινδύνους που δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Παραδείγματο χάρη, αυτή είναι μία εγκατάσταση σε μία σεισμογενή περιοχή και λέγεται ότι ε, δεν μπορεί να αντέξει σε περίπτωση σεισμού και δεν μπορούν να υπάρξουν και βελτιώσεις σε αυτή την κατασκευή. Εγώ, όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη χρηματοδότηση, ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, και τα θέματα ασφάλειας και την ασφάλεια της Λιθουανίας έναντι της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος Γιούροβα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε Ευχαριστώ κύριε Χάρμς για τα όσα είπατε σαν εισήγηση. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την έκθεση η οποία εγκρίθηκε στις 21 Δεκάτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε και για την ε, ε, ψηφοφορία που έγινε νωρίτερα σήμερα όσον αφορά την, ε, τις άλλες εγκαταστάσεις που όπως συναρμολογήθηκαν και όλα αυτά για τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους εμάς και το πόσο βοηθήσατε δείχνουν το πόσο ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει επομένω να έχουμε όσο γίνεται ψηλότερα πρότυπα ασφαλεία, διαφάνεια σε σχέση με κινδύνους σε σχέση με δαπάνε, σε σχέση με, με τον άμεσο παροπλισμό και δεν θα πρέπει να μετακυλίεται αυτό το βάρος στις επόμενες γενιές. Έτσι, έχουμε σημαντική μείωση όσον αφορά τον εθελοντικό κίνδυνο που τώρα έχει μειωθεί, ο κίνδυνος για, το γενικό, για τον κόσμο. Ε, και τώρα αυτά τα καύσιμα τώρα βγαίνουν από τον αντιδραστήρα και πηγαίνουν σε χώρους αποθήκευσης ασφαλής. Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί. Οπότε είχαμε αποσυναμολόγηση αυτών των εγκαταστάσεων και επίσης είχαμε την μεταχείριση, την δέουσα των αποβλήτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό, από το 2001, τα υποστηρίζει όλα αυτά οικονομικά και στην φάση της προένταξης ή στην Λιθουανία. Είχαμε ζητήσει από τη χώρα να κλείσει ε, τον σταθμό αυτόν που είναι του στυλ του Τσερνομπίλ, πιο μεγάλος και επίσης δώσαμε ενίσχυση οικονομική για να αντισταθμίσουμε την ε, ζημία. Είναι θέμα ελεγγύης το πώς θα αντισταθμίσουμε το κλείσιμο της Εγκυναλίνας στο τέλος του 2020 θα έχουμε δώσει 1,9 δις ευρώ οικονομική βοήθεια. Και προτείνουμε να συνεχιστεί η δέουσα βοήθεια στο μέλλον. Με αυτό το πρόγραμμα παροπλισμού θα αρχίσουμε να αποσανολογούμε τον πυρήνα του αντιδραστήρα έχει κάνει σχετικές προτάσεις στο Ελληνικό Συνέδριο. Έχουμε ένα το όριο συγχρηματοδότησης. Δεν θα υπάρχουν ε, ε, αμφισημίες και αμφιβολίες. Είναι το πρώτο στο είδος του αυτό το πρόγραμμα. Είναι διαστάσεων πρωτόγνωρων. Οι καλύτεροι ειδικοί έχουν εμπλακεί γιατί η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων είναι υψηλή προτεραιότητα. Επιστατεύσαμε την εμπειρία τους και ελπίζουμε ότι θα ωφεληθούν και άλλα προγράμματα έτσι. Και θα έχουμε έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ένωση. Θα πρέπει να μοιραστούμε τις ε, γνώσεις μας, θα πρέπει να έχουμε όσο μεγαλύτερη προσθέμενη αξία εις όφελος των ε, Ευρώπη. Ε, σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Και τώρα θα αρχίσουμε για τις, με τις παρεμβάσεις των ε, πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ. Κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ευχαριστώ την εισηγήτρια. Παλέψαμε πολύ για τη χρηματοδότηση Τελικά ε, συμφωνήσαμε μετά από πολλές διαφωνίες στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Η Λιθουανία χρειάζεται τη βοήθεια αυτή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στο πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης ε, είχαν δοθεί αυτές οι υποσχέσεις. Μας είπε η Επίτροπος ότι ήδη έχουν διατεθεί 1,9 δισεκατομμύρια, μιλάμε για άλλα 780 εκατομμύρια και ε, το κενό, το χρηματοδοτικό κενό είναι ακόμη άλλα 1,6 εκατομμύρια. Ποσά τα οποία πρέπει συνολικά να εκταμιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη Λιθουανία με οικονομικά αποδεκτούς όρους, αλλά θα πρέπει, κυρία Επίτροπε, να κατηγορήσω την Επιτροπή γιατί πρότεινε 550 εκατομμύρια, ενώ η Λιθουανία ζήτησε 780. Τελικά συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε για το ποσό που ζήτησε η Λιθουανία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να κάνει ένα σωστό υπολογισμό των πραγματικών αναγκών. Και την τονίζω αυτή τη συζήτηση, γιατί τελικά μιλήσαμε με τον Επίτροπο Έτιγκερ, με τον Υπουργό Ενέργεια τη Λιθουανία, με την εισηγήτρια και του κοιόδη εισηγητέ. Και μέχρι την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο έπρεπε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση που δεν την έχουμε ακόμη και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα, παρότι θα ψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Εκ μέρου ε, των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ε, Κολούμπα Σεφ για ένα λεπτό. Σεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση ζητά 80% ε, και εκφράζουμε 86% ε, ε, εκφράζουμε το αίτημα για 86%. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Χάρμς και τον κύριο Λάγκεν, διότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά μαζί και για το θέμα της Λιθουανίας και για τα θέματα που αφορά την Βουλγαρία, τη Σλοβακία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση για το κοινό κέντρο ερευνών ε, σχετικά με την ε, ε, γνώση, με τις γνώσεις σχετικά με την, τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών και τη διάδοση των γνώσεων αυτών είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το αίτημά μα για 780 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερο ποσό δηλαδή από αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή. Σε μερικά θέματα δεν μπορεί να υπάρχει συμβιβασμό. Για το ECR έχει τώρα τον λόγο ο κύριος Τόμας Εύσκη. Ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε αυτόν τον κανονισμό του Συμβουλίου σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα αρρωγής για τον παροπλισμό αυτού του πυρηνικού σταθμού. Εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερο πρόσφατα προς επίπεδα ασφαλείας τέλος πάντων, αυτό το χρειάζεται η Λιθουανία από πλευρά τη ασφαλεία. Επομένω, είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση, κυρίω λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα υπαριθμών 2 σοβιετικού τύπου όπως στο Τσερνομπίλ. Αυτό το πρόγραμμα όπου να είναι θα ολοκληρωθεί. Είπαμε τι θα γίνει με τον πυρήνα γραφίδι. Πολύ σημαντική αυτή η φάση και εάν δεν δοθούν τα χρήματα που χρειάζονται θα σταματήσει αυτή η αποσυναρμολόγηση. Ε, τότε θα τεθεί ένα αμφιβόλο υπόθεση ασφάλειας στην Ένωση. Η Λιθουανία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει όσο χρειάζεται την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν δαπάνες επιπλέον όσον αφορά τον παροπλισμό αυτού του σταθμού. Ο στόμας αυτός ήταν πάρα πολύ σημαντικό εργοδότης. Έχει υπάρξει σύγκριση του εισοδήματο και υπάρχει υψηλότερη ανεργία στη χώρα εκεί πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη χώρα. Οπότε θα πρέπει να δοθεί αυτή η δική χρηματοδοσία. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Για τους πρασίνους τώρα έχει τον λόγο ο κύριος Ρόπε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την αγαπητή συνάδελφο Ρεμπέκα Χάρμς από την ομάδα των Πρασίνων. Χαίρομαι που η έκθεση για το πυρηνικό σταθμό της Γναλίνα δόθηκε στην κυρία Χάρμς γιατί είναι από τους πιο ισχυρούς βουλευτές ε, για τα θέματα πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή συνεισφορά στο πρόγραμμα παροπλισμού θα πρέπει να είναι υψηλότερη με χαμηλότερη συμμετοχή της Λιθουανίας. Σήμερα συνεισφέρει κατά 14% η Λιθουανία και είναι τεράστιο χρηματοδοτικό βάρος για τη χώρα μου. Χαίρομαι που η Επιτροπή Ήτρε δέχθηκε την αύξηση της χρηματοδότησης και δέχθηκε να δοθούν και 200 εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι στην πρόταση της Επιτροπής για τον παροπλισμό. Η ψηλότερη χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται σε λεπτομερείς αξιολογήσεις που θα πρέπει να γίνονται από διεθνείς εμπειρογνώμονες. Εκτός από τα θέματα παροπλισμού, η Λιθουανία πρέπει να αντιμετωπίσει και τα δημογραφικά και κοινωνικά προβλήματα. Εγώ ήμουν δήμαρχος στην περιοχή του Ιγναλίνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χαίρομαι που η έκθεση αναφέρει τη δέσμευση της Λιθουανίας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανεργίας, έλλειψης εισοδημάτων και δημοσίων υπηρεσιών στην περιοχή. Τέλος, ευχηστώ την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι η ψηφοφορία αύριο θα δώσει ένα μήνυμα για το αν οι πολίτες θα δείχνουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκουόγκα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και σε όλη την ομάδα γιατί η ομαδική δουλειά ήταν πολύ σημαντική για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα και να αυξήσουμε το ποσό σε σχέση με αυτό το οποίο προσπάθησε να κόψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια χώρα που υποστηρίζει τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λιθουανία είναι η πιο ισχυρή υπέρμαχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α το λάβει υπόψη λοιπόν η Επιτροπή και α προσαρμόσει την χρηματοδότηση, ούτω ώστε αυτό ο αντιδραστήρα να κλείσει. Είναι εξίσου κακό αυτό ο αντιδραστήρα όπω και του Τσερνομπίλ που εξεράγει. α εξασφαλίσουμε λοιπόν τη χρηματοδότηση και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας βοηθήσει σε αυτό, διότι οι πολίτες πραγματικά ε, το περιμένουν αυτό. Το κλείσιμο του αντιδραστήρια δημιούργησε ε, προβλήματα και η χώρα χρηματοδότησε ε, τη διαδικασία αυτή σε μεγάλο βαθμό. Περιμένουμε τώρα ότι θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γουόγκα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπαλτσίτης για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες ε, προς την κυρία Χάρμς ε, και επίσης ε, και προς τον ε, σκιώδη συγητή, του συνάδελφό μου κύριο Κόρουμπας. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων ε, προς συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες που κατανόησαν την κατάστασή μας και μας στηρίζουν στο δύσκολο αυτό καθήκον στον παροπλισμό του πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο παροπλισμός αυτού του αντιδραστήρα δεν είναι μόνο μία πρόκληση για τη Λιθουανία, είναι ένα βάρο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πρέπει να αναλάβουμε αυτό το φορτίο γιατί θέλουμε την ασφάλεια. Οι Λιθουανοί εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενέκριναν ε, κάποιες δεσμεύσεις υπό το πρωτόκολλο 4 Γι' αυτό λοιπόν τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, αυτό θα σημαίνει ότι στρέφεται κατά των δεσμεύσεών της. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο ε, συμφωνεί με το να συγχρηματοδοτήσει ε, στην αποσυναρμολόγηση ενός από τους μεγαλύτερους αντιδραστήρες. Το λόγο έχει ο κύριος Ουροτσέφ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτόν τον κανονισμό και είναι σωστές οι τροπολογίες της κυρίας Χάρμς. Ο σκοπός είναι να συνεχιστεί η βοήθεια από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιγναλίνα να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση του παραπλησμού. Ε, ε, αυτά τα 700 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι επαρκή σχηματοδότηση για το πρόγραμμα και έτσι λαμβάνεται υπόψη αυτό το οποίο είπαν οι ειδικοί. Έτσι θα είμαστε πιστοί στο χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι δεν θα πρέπει να διακοπεί ε, αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι περίπλοκη. Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη αποσυνομολόγηση των μονάδων εκεί θα πρέπει να σταματήσουμε το ραδιολογικό κίνδυνο και δεν συμφωνούμε ότι μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση από το κράτος θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η σημερινή αναλογία συγχρηματοδότησης 86-14 δηλαδή και η αδίποτε αύξηση ε, της ε, αναλογίας εις βάρος του κράτους θα ήταν κάτι το αφόρητο από το κράτος θα ήταν πολύ βαρύ για τον κόσμο και αυτό θα μαύρωνε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ήταν διάψευση της υπόσχεσής της προς τους Λιθουανούς ευχαριστούμε συνάδελφε Γκρέσλε ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ. η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών επισκέφθηκε και, τους, και τα τρία, τους τρεις πυρηνικούς σταθμούς. Στο τέλος στην Ιγκλαλίνα τον Ιουνίου του 2018 πήγα δύο φορές. Κατανοώ ότι όλοι οι συνάδελφοι από αυτές τις χώρες προφανώς ενδιαφέρονται για περισσότερα χρήματα για την αποσυναρμολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απλούστευσε λιγάκι την όλη κατάσταση, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Το 2009 υπήρξε μία ε, διεθνής μελέτη σκοπιμότητας ε, για εναλλακτική αποσυναρμολόγηση αφού θα αφαιρεθούν οι ράβδοι του γραφίτη. Το 2010 μετά από πίεση των Λιθουανούν ε, ακυρώθηκε και έτσι λοιπόν το θέμα έκλεισε. Εκείνο το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο σταθμός Ιγκυναλίνα θα παραμείνει πυρηνικός. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να αναζητηθούν εναλλακτικέ λύσεις αντί για ένα πράσινο λιβάδι που δεν θα βοηθήσει κανέναν απολύτως. Πολύ ωραία. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία Catch the Eye. Ε, δύο ξεκινάω με τον κύριο Πόσπισιλ. Παρακαλώ. Πώς ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω μελετήσει το θέμα και θεωρώ, είμαι πεπισμένος ότι αυτά που ζητεί η χώρα είναι δικαιολογημένα, είναι βάσιμα. Θα πρέπει να συνεχιστεί το 14% ως συγχρηματοδότηση από τη Λιθανία. Αν το αυξήσουμε, τότε θα είναι πολύ άσχημη εικόνα που θα δώσουμε για την Ένωση και σε κάποιες χώρες που περάσει από τον κομμουνισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει και τόση δημοφιλία. Προσέχτε τις πολιτικές διαστάσεις του θέματος. Είναι πιο σημαντικό αυτό παρά αυτά τα 200 εκατομμύρια που θα κοπούν ή θα δοθούν παραπάνω. Άρα μην τα ξεχνάτε αυτά. Στη Λιθουανία ο κόσμος θα πρέπει να θεωρεί την Ένωση ε, σαν κάποιον που τηρεί τις υποσχέσεις του, να βοηθηθεί η Γκριναλίνα. σημαντικό το εγχείρημα να αποσυναρμολογηθεί ο πυρηνικός σταθμός στην Ινγκαλίνα διότι πρόκειται όπως υπόθηκε για παλαιούς αντιδραστήρες ίδιου τύπου με αυτό στο τσέρνομπιλ. άλλωστε κάτι τέτοιο έχει γίνει ήδη στην σλοβακία υπάρχει μια διαδικασία και για τον αντίστοιχο πυρηνικό σταθμό στη βουλγαρία στο κοσλοντούι όπου εκεί διαβάζω ότι η αποθήκευση των ραδιοενεργών υλικών θα γίνει στη βουλγαρία. το ερώτημα είναι τα ραδιοενεργά υλικά από την αποσύρμαν από τη διάλυση εν πάση περιπτώσει του σταθμού στη Λιθουανία πού θα αποθηκευτούν. Πού θα αποθηκευτούν τα ραδιενεργά απόβλητα. Μήπως στο Κόσοβο, μήπως στα Σκόπια. Θέλουμε μια απάντηση, διότι αυτό είναι επίσης σημαντικό, ο τρόπος στον οποίο θα αποθηκευτούν τα ραδιοενεργά απόβλητα από εκεί και πέρα συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της κυρίας harms και για υπάρχοντα πυρηνικά εργοστάσια να πω ότι είναι επικίνδυνο πλέον το εργοστάσιο το πυρηνικό που θα γίνει στο ακούγιο στην τουρκία. είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό η ευρωπαϊκή ένωση. μην εμφανιστούμε πάλι μετά από χρόνια εδώ και πληρώσει η ευρωπαϊκή ένωση το κόστος για την αποσυνορμολόγηση του πυρηνικού εργοστασίου στο ακούγιο. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε και δίνω το λόγο στην Επίτροπο, κυρία Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τα πολύτιμα σχόλιά σα. Από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει και υποστηρίζει τον παροπλισμό του Ιγναλίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, ε, όπως ε, παρατίθεται στην συνθήκη προσχώρησης της Λιθουανίας. Έχει συμφωνηθεί και από τη Λιθουανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προγραμματίζονται ε, οι διαδικασίες μέχρι το 2038, οπότε και θα έχουμε το οριστικό κλείσιμο και τα διεργά απόβλητα θα έχουν διατεθεί με σωστό τρόπο. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει όλες τις ανάγκες ε, για τις διαδικασίες μέχρι το, που θα ξεκινήσουν μέχρι το 2027. Όσον αφορά την έκκλησή σας για αύξηση του προϋπολογισμού, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα, δεν έχω την αρμοδιότητα από τους συναδέλφους, αλλά θα ενημερώσω το Σώμα των Επιτρόπων για το αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δέσμευσή τους για την πρόθεση του θέματος αυτού στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πακέτου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και δίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ρεμπέκα Χάρμς για την απάντησή της. Μία πρόταση μόνο προς τη συνάδελφο κυρία Γκρέσλε. πιο ασφαλής, ε, ε, πιο ασφαλές ε, κλείσιμο και αποξύλωση θα μπορούσε να είναι πολύ θετικό για μας, αλλά στην Γερμανία μπορεί να μιλάμε για οικολογικά μέτρα, αλλά σε άλλες χώρες μπορεί να καθυστερούν περισσότερο ε, οι διαδικασίες και στην ε, Λιθουανία πρέπει να προωθήσουμε την αποξήλωση. Όπως είπε ο κύριος Λάγγεν, είναι ε, μια αυθαίρετη αλλαγή στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα θέματα που ανέφερε η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση. Από τις επισκέψεις μου στη Λιθουανία κατέστησα σαφές ότι υπάρχει μια παραμέληση της Λιθουανίας και μια αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης της Λιθουανίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερο φταίει το Συμβούλιο γιατί δεν είναι η Επιτροπή η μόνη υπεύθυνη, είναι και το Συμβούλιο που θα πρέπει ε, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της Λιθουανίας στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους σκιώδεις συζητητές. Έκλεισε λοιπόν η συζήτηση και αύριο θα ψηφίσουμε. Σας ενημερώνω ότι αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσουμε στις 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 4 ε, ε, και μπορείτε να δείτε την ημερήσια διάταξη στην ιστοσελίδα. Λίγη τη συνεδρία.